και γίνεται ψηφοφορία αμέσως τώρα. Ξεκινούμε με τις ψηφοφορίες λοιπόν. Με πρώτο το θέμα της κατάστασης Ταϊλάνδη, μία ψηφοφορία για ένα ψήφισμα κοινό, πέντε ομάδων, χωρίς τροπολογίες. Τελική ψηφοφορία λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κοινό ψήφισμα πέντε ομάδων για το δικαίωμα στην εκπαίδευση στην υπερδνηστερία περιοχή. Έχουμε επιμέρους τροπολογίες παράγραφος 4 στο αρχικό κείμενο με προφορική τροπολογία του κύριου Μπρίντα. Παρακαλώ. Το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ θα πρότεινα στο τέλος του παραγράφου 4 να προσθέσουμε ε, ενημερώνοντας τις ε, πληροφορίες ε, και περιλαμβάνοντας και τις συλλήψεις ε, του γυμνασιάρχη και του λογιστή. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν. Τέταρτη παράγραφο, αυτή τη μορφή Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εννέα αρχικού κειμένου Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. τυολογική σκέψη α, δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά Αποχέ συγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά Αποχέ συγκρίνεται και αυτό λογική σκέψη γιώτα αρχικό κείμενο με τροπολογία προφορική του κυρίου Πρέντα e- Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση πρόκειται περί επικαιροποίηση των στοιχείων. Στο τέλος λοιπόν της τελική σκέψης να προσθέσουμε όσον ότι κρατήθηκαν ο λογιστής και η γυμνασία του Τσάντα Χάι όταν ε, μετέφεραν τους μισθούς ε, του προσωπικού. Αντιρρήσεις. Όχι, υπέρ παρακαλώ. Με τροποποιημένη μορφή. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη. Ο μικρόν αρχικό κείμενο, προφορική τροπολογία του κ. Ρεπ Ευχαριστώ. Μία τεχνική διευκρίνηση στην παράγραφο αυτή. Το Σεπτέμβριο του 2014 αναφερόταν όχι μετά τα τέλη Αυγούστου 2014. Μία μικρή αλλαγή. Ο Αύγουστος γίνεται Σεπτέμβριος. Γιατί έτσι γίνεται πιο συνεκτικό το ψήφισμά μας με το θέμα του Συμβουλίου του Εκπαιδευτικού. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν αντιρρήσει ω προ την προφορική τροπολογία. Όχι. Το ψηφίζουμε λοιπόν το κείμενο με τη μορφή αυτή. Υπάρχουν αντιρρήσει. Κύριε Πρέτο. Ε, δεν φτάνετε εσεί. Ψηφίζουμε την αιτιολογική σκέψη όμικρον με τη μορφή αυτή στο αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαληθεύουμε. Αιτιολογική σκέψη όμικρον. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. Το σύνολο της εκθέσεως, της, ε, ψηφίσματος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τελευταία ψηφοφορία για σήμερα το ψήφισμα για τον Μπαχρέιν και ιδιαίτερα τι περιπτώσεις Ναμπίλ Ρατζάπ, Απτουλ Αλκαουάια και Ιμπραήμ Σαρίφ. Πρόταση ψηφίσματο τεσσάρων ομάδων και τι τροπολογίε παράγραφος 8, αρχικό κείμενο πρώτο κομμάτι, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται παράγραφος 8 Τρίτη, πρώτη τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. σε 9, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. παράφος 10, αρχικού κειμένου, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Μετά την παράγραφο 14, τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. με 7 αποχές, 48 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο καλά, ε, κατά. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επάνωδο. Ο κύριος Οντί όμως για το διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, ζήτησα το λόγο προηγουμένως όταν ε, ψηφίζαμε την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου όσον αφορά το οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσαρμογή των προσωστώσεων ε, εκπομπών του ανθρώπου, Δεν μου δόθηκε ο λόγος και να υπενθυμίσω τον κανονισμό για την πολυγλωσία, διότι ψηφίσαμε τη θέση του Κοινοβουλίου και ο κανονισμός επί του οποίου ψηφίσαμε από τη μία πλευρά δεν εμφανίζεται στη σελίδα του Seance on Direct και δεν έχει μεταφραστεί. Λοιπόν, οι βουλευτές ψήφισαν ένα έγγραφο που, που παραβίαζε τους κανόνες περί πολυγλωσίας. Είναι μια νέα απόπειρα για την ε, μείωση της πολυγλωσίας ε, στο Κοινοβούλιο. Μιλάω για την Ολομέλεια, δεν μιλάω για τις Επιτροπές. Θα ήθελα λοιπόν να κάνετε μια παρατήρηση προς την Προεδρία, ώστε η πολυγλωσία να πάψει να υποβαθμίζεται στο Ευρωπαϊκό μας Κοινοβούλιο.